Uh, Συνάδελφοι, κύριε και κύριοι, περίμενα λίγο γιατί ξέρω ότι δεν ήταν καλά τα πράγματα στους δρόμους, είχε πολύ ποτηλιάρισμα, αλλά παρόλα αυτά λέω να ξεκινήσουμε, να μην καθυστερήσουμε άλλο. Και γυρνάω στα γερμανικά. Θέλω λοιπόν να σας ε, καλωσορίσω στην πρώτη συνεδρίασή μας για φέτος. Χαίρομαι που σας βλέπω, σας εύχομαι κάθε ευτυχία για το 2020. Εισαγωγικά να πω, θα ξαναγυρίσω στα αγγλικά και για λόγους ευγένεια για τους ε, συναδέλφους μας από, την, ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο. Συνάδελφοι, ε, σήμερα είναι σχεδόν σίγουρα η τελευταία φορά που έχουμε μαζί μας τους Βρετανούς συναδέλφους μας εδώ σε συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμότατα όλους για τη σκληρή σας δουλειά, για την αφοσίωσή σας Κάποιοι από εσά, όπω η Τζούλι Γουόρντ, ε, είστε μέλη τη Επιτροπή Κούλτ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άλλοι είναι πιο νέοι από την αρχή τη κοινοβουλευτική περίοδου αυτή που διανύουμε. Αλλά είναι μια περίεργη ημέρα, είμαι βέβαιη για όλου σα. Περίεργε εβδομάδε. Τελειώνει η θητεία σα, η κοινοβουλευτική, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ λυπημένη που σας βλέπω να φεύγετε. Χαίρομαι όμως που είχαμε την ευκαιρία να ε, δουλέψουμε μαζί τους τελευταίους μήνες και χρόνια. Το πάθος σας για την παιδεία και τον πολιτισμό, η προσήλωσή σας στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και η σκληρή σας δουλειά θα μας λείψει. Εκ μέρου ε, τη Επιτροπή Παιδεία και Πολιτισμού θέλω να σα ευχηθώ ό,τι καλύτερο για το μέλλον και να σα ξαναευχαριστήσω για τη δουλειά σα. σω δε υπάρξουν και κάποιε νέε ευκαιρίε για Όπω και αν διαμορφωθεί η μελλοντική συνεργασία μεταξύ Βρετανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. επομένω ίσως σε άλλους ρόλους, με άλλες ιδιότητες, να ξανασυναντηθούμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ για, την, για την δουλειά σας, τη συνεργασία σας. Εγώ θα ήθελα να είχατε μείνει. Διαφορετική ήταν όμως η απόφαση που ελήφθη. Σας ε, εύχομαι λοιπόν ε, καλό δρόμο και ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις από πλευρά σας, εγκρίνεται η σε διάταξη με τη μορφή που έχει. Υπάρχουν αντιρρήσεις ή ενστάσεις. Όχι. Το σχέδιο πρακτικών της συνεδρίασης της 4ης Δεκεμβρίου το έχετε λάβει στα έγγραφα της συνεδρίασης. Υπάρχουν παρατηρήσεις όσον αφορά τα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής. Όχι. Ωραία. Άρα θα θεωρηθεί ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί σε περίπτωση που δεν υποβληθούν ενστάσεις ή αντιρρήσεις στη διάρκεια της ε, συνεδρίασής μας. Για τη διερμηνία. Έχουμε διερμηνία σήμερα σε εξή γλώσσες, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, ουγγρικά, λετονικά, πολωνικά, σλοβακικά, σλοβενικά, βουλγαρικά, ρουμανικά και κροατικά καλύπτουμε όλες τις γλώσσες των ε, παρισταμένων. Βλέπω ότι κάποιος ζητά το λόγο. Παρακαλώ. Mm, κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα απλώς να ε, προσθέσω στα εισαγωγικά σας σχόλια και να σας πω πως η κυρία Νόμικα Σεμέντο θα είναι η αντικαταστάτρια στην Επιτροπή Πολιτισμού και η οποία είναι μέλος, ε, πλήρες μέλος στην ε, Επιτροπή ε, Απασχόλησης. Σας την συστήνω σήμερα γιατί θα είναι η νέα μας εκπρόσωπος, αναπληρώτρια. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Σας καλωσορίζουμε και προσβλέπουμε σε μια καλή συνεργασία τα επόμενα χρόνια μαζί σας. Ευχαριστώ, λέει η κυρία Σεμέντο. Τζούλη. Ευχαριστώ και για τα καλά σου λόγια, Σαμπίνε. Δεν θέλω να απαντήσω, να σου πω την αλήθεια, γιατί είναι πολύ συναισθηματική στιγμή για όλους μας. Ε, είμαστε εδώ γιατί μας νοιάζει. Αυτοί που δεν τους νοιάζει ε, δεν είναι εδώ σήμερα και δεν ήταν και ποτέ όταν χρειαζόταν. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έφερα σήμερα μαζί μου έναν νεαρό ε, πολιτιστικό ηγέτη είναι εδώ μαζί μου και θέλω να τον χαιρετήσω γιατί ο πολιτισμός ε, και η νεολαία είναι το μέλλον. Θέλω λοιπόν να σας ε, παρουσιάσω τον Μάθιο που κάθεται εκεί πίσω. Το μέλλον είναι η γενιά σου. Είμαι βέβαιη ότι το ενδιαφέρον του για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και η ενέργεια του, το πάθος του θα εξασφαλίσουν ότι στο μέλλον οι νέοι άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο θα, είναι, θα συνεχίσουν να είναι συνδεδεμένοι. Είναι μέλος ε, του προγράμματος ΚΛΟ που είναι ένα πρωτοπόρο ε, πρόγραμμα στην Βρετανία για νέους ανθρώπους και τον πολιτισμό. Ευχαριστώ λέει Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ Τζούλη που φέρνεις και νέους ανθρώπους γιατί είναι πραγματικά σημαντικό να έχουμε νέους ανθρώπους ηγέτες από τη Βρετανία που θα μείνουν σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ε, γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα που δυστυχώς δημιουργήθηκε από τον Brexit. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας. Λοιπόν, Επιστρέφω στις ανακοινώσεις μου. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε κόσμοι εδώ μέσα. Προφανώς μας βλέπουν αποφάσεις ε, των συντονιστών της 4ης ε, Δεκεμβρίου 2019 να σας ανακοινώσω ότι οι αποφάσεις των συντονιστών της 4ης Δεκεμβρίου που απεστάλησαν στις 6 Δεκεμβρίου στα μέλη της ε, Επιτροπής Κούλτ έχουν εγκριθεί καθώς δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις έως την προθεσμία που είχε οριστεί την 9η δηλαδή Δεκεμβρίου. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρας διάταξης Σχέδιο γνωμοδότησης, απαλλαγή 2018, Γενικός Προπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ηλεκτρονική ψηφοφορία και μετά θα γίνει και μια ψηφοφορία για το Μεταφραστικό Κέντρο. Εγώ είμαι συντάκτρια της, ε, γνωμοδότηση ε, της γνωμοδότησης και θέλω να σας ε, ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω τους σκιώδεις με τους οποίους συνεργαστήκαμε, όλα τα μέλη της Επιτροπής που υπέβαλαν τροπολογίες Οπότε νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις ε, ηλεκτρονικές σας κάρτες μαζί, τις κάρτες ψηφοφορία. Από τεχνική απόψεως λειτουργούν όλα καλά. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν με την ε, ε Γενική Απαλλαγή 2008, Απαλλαγή 2008 Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάμε. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 4 αποσύρθηκε. Περνάμε στην τροπολογία 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Όχι, συγγνώμη. 6. 6. Ε, γιατί καταπίπτουν 3 και 19. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18. Με προφορική τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε σας παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα της ψηφοφορία λοιπόν. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε και εγκρίνεται με μεγάλη πλειοψηφία. 24 υπέρ, 3 κατά, μία αποχή. Και περνάμε στο επόμενο θέμα, απαλλαγή του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένωση. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ κατά, αποχές, όχι σε δύο τμήματα, συγγνώμη. Λοιπόν, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία και πάλι ηλεκτρονικά. Ψηφίστε σας παρακαλώ με τις κάρτες σας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. 27 υπέρ, μία αποχή, εγκρίνεται και αυτή η γνωμοδότηση με μεγάλη πλειοψηφία. Σχεδόν ομόφωνα. Σας ευχαριστώ λοιπόν και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 7. Στρατηγικό θεματολογίο καινοτομία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομία και Τεχνολογία, τόνωση του αλέντου και τη ικανότητα για καινοτομία τη Ευρώπη. Συντάκτρια τη γνωμοδότηση είναι η Judith Bunting. Καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή Ήτρε. Πρωτού δώσω το λόγο σε συντάκτρια της γνωμοδότηση, θέλω να σας ενημερώσω ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι στις 27 Ιανουαρίου στις 4 ώρα το απόγευμα και η ψηφοφορία στην Επιτροπή θα γίνει στις 17 Μαρτίου. Να δώσω το λόγο στην κυρία Μπάντινγκ. Παρακαλώ. Hello, um... Γεια σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και ευχαριστώ για τα αρχικά σχόλια. Παρακαλώ όσοι αποχωρείτε την αίθουσα, με ησυχία σας παρακαλώ, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους για τις ευχές τους εν ώψη του Brexit. Πραγματικά είναι κάτι φρικτό. Να πω ότι αισθάνομαι προνομιούχα που είχα τη δυνατότητα να συμμετάσχω σε ένα τέτοιο θέμα τόσο κοντά στην προθεσμία βέβαια, στην καταληκτική. Η έκθεσή μου αφορά τη στατική ατζέντα καινοτομία για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Είναι κάτι που δεν το είχα ξανακούσει μέχρι που ανέλαβα το θέμα. Γιατί το λέω. Πέρα από την ένθερμη υποστήριξή μου για την παιδεία και γι' αυτό είμαι σε αυτή την επιτροπή, Ήμουν και δημοσιογράφος για 30 χρόνια και με απασχολούσε αυτό το θέμα όταν κατάλαβα αυτό το ίδρυμα υπήρχε και δεν το είχα ακούσει ποτέ. Συγχωρέστε με. Ρώτησα διάφορου συναδέλφου τη Επιτροπή Κουλτ και διαφόρου στην αντιπροσωπεία μου και πολλοί ευρωβουλευτέ δεν το ξέρουν αυτό το κέντρο τη ε, καινοτομία. Παρακαλώ να έχετε υπομονή να μιλήσω πρώτα απ' όλα για αυτό το φορέα πριν αναφερθώ στην ε, νομοθεσία. Καταρχά, το 2019 τον Ιούλιο που μας πέρασε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα νέο νομοθετικό πακέτο. Συμπεριλαμβάνει αναδιατύπωση, που ο Κριστιαν Έλλαρ θα το αναφέρει αυτό αργότερα, και το θεματολόγιο για την καινοτομία δική μου ευθύνη και έχει παράρτημα 27 σελίδων το κείμενο, η δέσμη αυτή. Το πακέτο καθορίζει την ατζέντα και τον προπολογισμό για την επόμενη επταετία και εμείς σαν Επιτροπή δίνουμε στο κέντρο τεχνολογίας 3 δις ευρώ για να εργάζεται. Και αυτά τα ευρώ δαπανώνται σε όλη την Ευρώπη προς υποστήριξη της παιδείας, της έρευνας και των επιχειρήσεων. Και έτσι το EIT είναι ενδιαφέρον. Δεν είναι απλώς ακαδημαϊκό ίδρυμα, είναι ένα στεσμός που έχει σχεδιαστεί με την πρόθεση να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, την εμπορική ανάπτυξη. Ποια είναι η ιδέα. Αν ενθαρρύνουμε την καινοτομία, ή αν δημιουργηθεί καλό κλίμα για καλή τεχνική ε, καινοτομία, να έχουμε την παιδεία που υποστηρίζει όλα αυτά και αν έχουμε επικεφαλή επιχειρήσεων που ξέρουν πώς να εμπορευματοποιήσουν νέες ιδέες και υπηρεσίες, μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης. Από θέσεις απασχόλησης παίρνουμε φόρους, αν τι επιτυχείς επιχειρήσεις έχουμε φόρους λοιπόν, υπηρεσίες και έχουμε μια βιώσιμη οικονομία. Πολλά συμπεριλαμβάνονται αυτή την νομοθεσία, τα οποία θα επεκτείνουν την εμβέλεια του Ιδρύματος πέρα από τους κεντρικούς φορείς και τις βασικές επιχειρήσεις. Θα ακούσετε περισσότερα από τον Κρίστιαν. Και εγώ θα μιλήσω γι' αυτά όμως. Γιατί δεν το έχουμε ακούσει το Ίδρυμα αυτό. Είναι ένας καλός οργανισμός Ανησύχησα, ανησυχούσα αρχικά για την ποιότητα της έρευνας, αλλά από ό,τι έμαθα μέσω των ενημερώσεων που είχα, ήταν ότι το EIT έχει κάνει έξοχη δουλειά και έχει μια πολύ καλή ιστοσελίδα, αλλά πρέπει να εστιαστούμε επί της ε, εμπορικής πρόθεσης των υπηρεσιών. Θα έπρεπε να ξέρουμε τι κάνει αυτό το Ίδρυμα στην περιοχή μας για την παιδεία, πια για την ευρωπαϊκή βιώσιμη ανάπτυξη. Ο θεσμός αυτός δεν έχει τη μορφή κανονικού ε, πανεπιστημίου. Δεν έχουμε μια κεντρική μονάδα που γίνεται η έρευνα, έχουμε ένα διοικητικό κέντρο και από εκεί ε, ξεκινά ένα συστός, ένα δίκτυο διαφόρων φορέων και επιχειρήσεων που συνεργάζονται. Και έτσι κατάφεραν να επεκταθούν σε όλη την Ευρώπη. Το EIT καλύπτει οκτώ τομείς. Τους θεωρώ σαν τμήματα, αποκαλούνται κοινότητες γνώσεως και κοινοτομίας. KRC. Ας πούμε ότι είναι τμήματα πανεπιστημίου, σχολές πανεπιστημίου. Καλύπτουν τμήματα όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι Ευρωβουλευτές κατά το παρελθόν θεωρούσαν ότι είχαν κάποια προβλήματα κοινωνικά, ενδεχομένω. Υγεία, Φερρυπίν, κλίμα, ψηφιακό τομέα, ε, διατροφή, ε, παραγωγή προϊόντων, αστικέ ε, μετακινήσεις, πρώτε ύλε. κάτι μου ξέφυγε. Μπορείτε να το δείτε στην ιστοσελίδα. Είναι κοινότητε γνώσης και καινοτομία. Και εκεί έχουμε διάφορα Ινστιτούτα, φορείς έρευνας και επιχειρήσει που συμμετέχουν, ιδιωτικέ και μεγάλες και μικρές επιχειρήσει και όλοι κινούνται σε αυτό το υπέροχο τρίγωνο της γνώσης που είναι και η ραχοκοκαλιά του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος αυτού, της τεχνολογίας. Έρευνα. Έχουμε ένα σύντομο έγγραφο για την καινοτομία με ένα παράρτημα 27 σελίδων. Έξοχο παράρτημα. Και ένα από τα πράγματα που προσπάθησα να κάνω είναι να δώσω μια γεύση από το παράρτημα και τις εξηγήσει που δίνει το παράρτημα και όλα αυτά τι εξηγήσει να τα εντάξω τι λεπτομέρειε στην νομοθεσία. Προτείνω 95 τροπολογίε. Ακούγονται πολλέ για γνωμοδότηση, αλλά δεν είναι, κατά την άποψή μου, είχα προσέξει στο παράρτημα. Αναφέρω νομικά στοιχεία. Από το παράρτημα τα φέρνω στο κείμενο, το διατακτικό. Κάποιε πληροφορίε πρέπει να αναφέρονται στο νομοθετικό πρόγραμμα αυτό καθεαυτό. αυτό. Οι τροπολογίε αφορούν γενικού γενικούς και ειδικού στόχου του EIT, προτεραιότητες για την κοινότητα γνώσης και καινοτομίας. Οκτώ τομείς. Να ξεκινήσει ένα τέτοιο νέο τομέα που αφορά το δημιουργικό τομέα και τον πολιτισμό. Προπολογισμό και συνεργασία με άλλα προγράμματα. Το EIT τροφοδοτείται οικονομικά από το πρόγραμμα Horizon. Μετά έχουμε το EIC, έχουμε καινοτομία, έχουμε διάφορα τμήματα του Ορίζοντα Ευρώπη και του Ορίζοντα 2020 και συνεργάζεται το Ευρωπαϊκό Αυτό Ίδρυμα Τεχνολογίας και Καινοτομίας με τους άλλους φορείς. Εντός της νομοθεσίας και του παραρτήματος γινόταν λόγος για την εκπαίδευση των επιχειρηματιών. Αυτό είναι καλό και αναγκαίο στοιχείο. Ένας από τους λόγους που αναφέρεται εκτενώς είναι γιατί έγινε ένα έλεγχο πριν από κάποια χρόνια που είπαν ότι δεν γίνονται αρκετά σε αυτόν τον τομέα στο EIT και όπως πάντοτε γίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το παρατράβηξε το σκηνή, το εκρεμές πήγε από την άλλη πλευρά προς τις επιχειρήσεις. Δεν θέλω να μειώσω αυτές τις προθέσεις, αλλά ήθελα να επαναφέρω την επιστήμη και τεχνική εκπαίδευση. Αν δεν έχει τεχνική παιδεία, και καλές τεχνικές ιδέες, τότε δεν έχεις επιχειρήσεις προς ανάπτυξη. Ακόμα και αν δεις τις υπηρεσίες, όπου εκεί εστιάζεται και το θέμα του κλίματος, χρειάζεται επιστημονική κατανόηση για την πρόθεση των διαφορών μέτρων. Οι τροπολογίες μου αφορούν και τη φιλοδοξία. Θέλω να είμαι σίγουρη ότι υπάρχει φιλοδοξία. Δεν πάει κατακτήσει τον κόσμο χωρίς φιλοδοξία. Ήμουν ήδη σε μια ενημέρωση τη υπηρεσία έρευνα που έλεγε ότι έχουμε μείνει πολύ πίσω στην Ευρώπη όσον αφορά την αποθήκευση ενέργεια, που θα μπορούσαμε να καταπαρατήσουμε. Εκεί να ηγείται. Θα έπρεπε να αστιαστούμε αλλού. Δεν το θέλουμε αυτό να μας δίνεται σαν συμβουλή για κανέναν άλλο τομέα εμπορίου και επιστημονικής ανάπτυξης, άρα χρειάζεται φιλοδοξία και θα δείτε πολλά φιλόδοξα στοιχεία στις Προείπα ότι, προανέφερα ότι ελάχιστα ακούσαμε για το EIT. Υποστηρίζω λοιπόν τον προπολογισμό για προώθηση εμπορική και ενημέρωση. Και έχουμε και ένα πρόγραμμα για περιφερειακή επένδυση που θα διαδώσει τα ωφέλη σε όλη την Ευρώπη, ούτω ώστε τα πιο καινούργια κράτη-μέλη να ωφεληθούν και αυτά. Και είναι κάτι που το υποστηρίζω μέσω τροπολογιών. Και ενέταξα κάποιε τροπολογίες για να εγγυηθούμε κάποια ισορροπία ε, των δύο φύλων και να δοθεί και η διάσταση του φύλου στα διάφορα μέτρα. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση για περαιτέρω διαφάνεια όσον αφορά τον τρόπο που λειτουργεί το EIT και τα διάφορα τμήματά του και αυτό διότι θεωρείται ότι εκείνοι που ήδη έχουν πάρει τα χρήματα, κρατάνε τους πόρους για αυτούς, χρειάζεται διαφάνεια του πώς ανατίθενται οι συμβάσεις και πρέπει να καθίσταται σαφές ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ευπρόσδεκτες. Αναφέρονται κάποιες ιδέες μετά που συζήτησα με το διευθυντή του EIT, είχα τι ιδέε. Αυτά θα προωθήσουν τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα είναι δυνατόν και ε, οικονομικά να συμμετέχουν οι μικρέ επιχειρήσει. Και έχουμε ένα νέο τομέα που προτείνουμε, ένα νέο τμήμα που θα καλύπτει τι δημιουργικέ ε, επιχειρήσει. Ξέρουμε ότι είναι μεγάλοι εργοδότε, ότι υπάρχουν λαμπρέ ιδέε στην Ευρώπη στον τομέα το δημιουργικό. Και εδώ η Ευρώπη, εμεί, εμείς ο πολιτισμικός τομέας μπορούμε να ωφελήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, έχετε τη γνωμοδότησή μου μπροστά σα. Ελπίζω να θέλετε να υποστηρίξετε τι τοπολογίε. Η προθεσμία είναι 27, λέτε, 27 του μηνό Μπορώ να ακούσω ερωτήσει σας και ευχαριστώ που με ακούσατε. Ε, να διορθώσω. 17. Όχι 27. Όχι, όχι. Εγώ έκανα λόγο. Όχι, έχετε, έχετε δίκιο. Πράγμα, πράγματι, 27 Ιανουαρίου. Σωστά τα είπατε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Αποσύρω. Σκιώδη. Κριστιαν Έλα. Έχει πρώτο το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις προσπάθειες που κάνατε. Ήμουνα 15 χρόνια εισηγητής για τα προγράμματα ε, πλαίσιο και τα προγράμματα ε, του ε, Horizon και θα ήθελα να προσθέσω και να απευθύνω μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τους πω το γεγονός πως το μέσο αυτό και το ίδρυμα αυτό δεν είναι τόσο γνωστό στο ευρύτερο κοινό, ε, ουσιαστικά προέρχεται από μια εσωτερική αντίφαση μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ήταν υπεύθυνε δύο ε, γενικές διευθύνσεις, είχε να κάνει με, οργανωτικά, με οργανωτικούς λόγους και όχι πολιτικούς, ε, και δεν προωθήθηκε επαρκώς το ίδρυμα αυτό, το Ινστιτούτο αυτό. Ξέρετε πως τα θέματα περιβάλλοντος, τα θέματα ε, αποθήκευσης ενέργειας ε, ήταν σε άλλες προσκλήσεις και 4 δις ευρώ δαπανήθηκαν για τις ευφυγείς πόλεις ε, το τελευταίο διάστημα χωρίς να υπάρχει καμία υποχρέωση ετούντες να ε, εντάξουν τα EIT, ε τα οποία βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη. Αλλά αυτά περιμένουν από εμάς ε, για να μπουν στο παιχνίδι και δεν καταλαβαίνουν ακριβώς πώς θα μπορούσαν να ενισχυθούν, να ενταχθούν στις ευρύτερες πολιτικές, να δραστηριοποιηθούν. Όταν λοιπόν αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να προωθήσουμε το εργαλείο αυτό, τότε πιστεύω πως θα πρέπει να ξεκινήσουμε προωθώντας το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο και θα πρέπει στις ευρύτερε ευρωπαϊκές πολιτικές να το εντάξουμε καλύτερα. Είτε ε, επειδή θα πιέσουμε εμείς, είτε ε, επειδή θα το κάνει η ίδια Επιτροπή. Αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά έχουμε ένα ίδρυμα, το και το οποίο ε, δραστηριοποιείται στο Ισραήλ στα προγράμματα που ε, ε, έχουμε στήσει εκεί. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αλλού. Θα μπορούσε να γίνει, για παράδειγμα, στο Μαρόκο, στις ε, χώρες, στο πρόγραμμα γειτονία στην Ευρώπη. Άρα, λοιπόν, θα πρέπει να εξετάσουμε πώς μπορούμε αυτό το Ινστιτούτο να ενταχθεί καλύτερα σε όλα τα επενδυτικά και χρηματοδοτικά σχήματα στην Ευρώπη Και έτσι θα, θα χρειάζεται τόση συζήτηση για τον προπολογισμό και τι δράσει ε, του Ινστιτούτου. Μ' αρέσει πάντω αυτό που έκανε η συγγήτρια. Νομίζω πω είναι η σωστή. Ε, η τακτική Καταλαβαίνετε βέβαια πως μεταξύ Ήτρε και Κάλτ εγώ κάπου αισθάνομαι ε, μια εσωτερική διαιρεση Ας το δούμε. Πιστεύω πάντως πως ε, το κομμάτι το εκπαιδευτικό το έχουμε υποτιμήσει. Και ε, επιχειρηματική εκπαίδευση που θα προσφέρουμε μέσω πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αν τα καταφέρουμε, γιατί οι δραπαγματεύσεις δεν θα είναι απλές, αλλά ίσως θα καταφέρουμε να υψώσουμε ε, τη φωνή μας και να τα πούμε όλοι ενωμένοι. Στο παρελθόν ε, δεν το έχουμε καταφέρει και ίσως θα πρέπει μαζί με την Κομισιό να πούμε αντί να περικόψετε τμήματα του προγράμματος γιατί αποτελούσε τον αποδιοπομπαίο τράγο να κάνουμε καλύτερες ε, προτάσεις γιατί ίσως είναι η πρώτη ευκαιρία αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει το ρόλο του τίμιου διαμεσολαβητή ε, στις προτάσεις για τον καινούργιο προϋπολογισμό και να μην είναι μία μάχη μεταξύ θεσμών οι οποίες ε, πολλές συχνά έχουν αποδυναμώσει το, τη θέση του Ινστιτούτου ε, στα πλαίσια των συζητήσεων και διαπραγματεύσεων που γίνονται για τον προπολογισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Ντομινίκ Ρόβις είναι ε, επόμενη ε, επόμενος αλλά δεν είναι εδώ. Η Τάτ Μελμπάντα έχει, τον, ε, έχει τον λόγο. Ε, thank you, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχήν να ξεκινήσω, την κυρία να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Μπάντινγκ που ήταν η συγγήτρια και έκανε πολύ καλή δουλειά έτσι ώστε να εγκρίνουμε τον φάκελο. Ο αριθμός τροπολογιών που ήταν σχεδόν 100 νομίζω αποδεικνύει πόσο δύσκολο ήταν και πραγματικά ευχαριστώ την εισηγήτρια για το γεγονός του ότι έδωσε ε, περισσότερη ε, σημασία στο θέμα ε, αυτό των πολιτιστικών ε, ιδρυμάτων. Πιστεύω πως θα χρειαστεί να ε, στηρίξουμε την καινοτομία στον τομέα των πολιτιστικό και των οπτικο-ακουστικό και να ξέρουμε πως οι άνθρωποι που καινοτομούν έχουν τις επιχειρηματικές γνώσεις για να ε, κεφαλαιοποιήσουν ε, αυτήν ακριβώς την τεχνογνωσία τους. Τώρα, για το σχέδιο ε, που προτείνεται, θα θέλαμε η επιλεξιμότητα να είναι καλύτερα εστιασμένη. Ξέρετε πως ο κατάλογος ε, για τους ε, ε, καινοτόμου μικρού μεγέθους συμπεριλαμβάνει όχι μόνο την Ανατολική Ευρώπη, αλλά την Ιταλία, την Ισπανία. Δηλαδή 40% της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που κάνει έρευνα και καινοτομία προέρχεται από επιλέξιμε χώρες. Μην ξεχνάτε πως η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη και γι' αυτό ζητώ η επιλεξιμότητα να βασίζεται στο κατάλογο χωρών που έχουμε στο Horizon Επίσης, για τα περιφερειακά σχέδια, ε, τα επενδυτικά, νομίζω θα πρέπει να περιορίσουμε το ποσοστό και να εξασφαλίσουμε πως θα υπάρχει και γεωγραφική ισορροπία. Όταν μιλάμε για γεωγραφική υπηρεσία και μιλάμε για συστεγασμένα ιδρύματα, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γίνεται να έχουμε πάνω από 10 ε, που να αποτελούν ένα κέντρο και για τα κέντρα αυτά, ο στόχος του Ινστιτούτου θα πρέπει να είναι να επιδιώκουν την οικονομική σταθερότητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτά τα κέντρα να έχουν και κάποιες στρατηγικές που να αποφέρουν έσοδα και για να εντάξουμε τις προτεραιότητες αυτές εγώ θα καταθέσω μια σειρά τροπολογιών και σίγουρα θα βρούμε κοινό τόπο εμείς και η εισηγήτρια και με χαρά περιμένω τις συζητήσεις που θα κάνουμε σχετικά. Äh, äh, Ευχαριστώ πολύ. Επειδή δεν έχουμε άλλον σκιώδη από κάποια άλλη πολιτική ομάδα μαζί μας, δίνω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας. Θέλει κάποιος να τοποθετηθεί? Όχι. Να ζητήσω λοιπόν από την εκπρόσωπο της Κομισιόν να, να παρέμβει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θετικά σχόλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τα σχόλια. Συναδέλφου Μπάντινγκ. Και όσα είπαν και οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές. Ευπρόσδεκτη η έμφαση στην παιδεία και την κατάρτιση. Και όπως αναφέρθηκε, η εκπαίδευση του, των επιχειρηματιών είναι κάτι που λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη, όπως και άλλα στοιχεία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι πρέπει να προωθηθεί αυτός ο τομέας, διότι είναι η καλύτερη δυνατή δράση. Να έχουμε υπόψη επίσης και τον αυτόνομο των διαφόρων τομέων του Ινστιτούτου. Προφανώς θέλουμε να συμμετέχουν περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις δραστηριότητες, όμως θα πρέπει οι δράσεις να κατευθύνονται, ούτω ώστε να καταλήξουμε στην οικονομική βιωσιμότητα που αναφέρθηκε ως σημαντικότατη ευπρόσδεκτική υποστήριξη στο νέο τμήμα για τις πολιτισμικές και δημιουργικές ε, ε, επιχειρήσεις. Είναι κάτι που στηρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προσβλέπουμε σε συνεργασία γι' αυτό. Το μόνο θέμα που θέλουμε να θίξουμε σαν πρόβλημα τις τροπολογίες προτείνουν το, μέχρι το 2028. Αυτό είναι εκτός του παρόντος δημοσιονομικού πλαισίου και θα πρέπει να βάλουμε το όριο πιο κοντά εντός του δημοσιονομικού πλαισίου. Να εξασφαλίσουμε επίσης ότι υπάρχει συνοχή μεταξύ των νομοθετικών προτάσεων και οι στόχοι θα πρέπει να εντάσσονται στην κοινή συνεννόηση στην οποία καταλήξαμε τον, στις 27 Μαρτίου για τον ορίζοντα Ευρώπη. Πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα χαράς ακούσαμε αυτές τις απαντήσεις και αυτά τα σχόλια από εσά. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Δεν βλέπω να υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Ο Κρίστιαν Έλα είναι ε, εισηγητής Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομία και Τεχνολογία. Αναδιατύπωση πρόκειται για μια γνωμοδότηση την οποία συνέταξε, οπότε δίνω κατευθείαν το λόγο στον Κρίστιαν Έλλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευπρόσδεκτη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όμως λείπουν λεπτομέρειες και λογική σαφήνεια και αυτή η αναδιατύπωση ίσως να ήταν η καλύτερη προσέγγιση. Προτείνω, για, προτείνω διάφορες τροπολογίες για μεγαλύτερη σαφήνεια νομική και να δοθεί και μια ασφάλεια δικαίου στον κανονισμό. Τα βασικά στοιχεία του κειμένου είναι εξασφαλιστή η χρηματοδότηση του ΙΕΤ με 4% του γενικού προπολογισμού του ορίζοντα Ευρώπη, όπως υθετήθηκε από το Ευρωκοινοβούλιο. Δεύτερον, να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένας τομέας για τον πολιτισμό και το δημιουργικό τομέα στο ΙΕΤ για την περίοδο 2021 μέχρι 2027 να εξασφαλίσουμε επαρκή χρηματοδότηση για την δημιουργία του τομέα χωρίς να υπονομεύεται η οικονομική βιωσιμότητα των υφισταμένων τμήματων του Ινστιτούτου. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε τα πάντα βέβαια στα τυφλά. Η οικονομική βιωσιμότητα δεν είναι μόνο υποχρέωση στο EIT που αφορά τον προπολογισμό και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι και υποχρέωση των διαφόρων τμήματων και τομέων του Ευρωπαϊκού Αυτοινστιτούτου. Δεν θα πρέπει τυφλά να υποστηρίζουμε τα πάντα. Καταρχήν όμως δεν πρέπει να υπονομεύουμε τα εφιστάμενα τμήματα. Ο εισηγητής θέλει να τονίσει ότι η προσπάθεια και έρευνα πρέπει να αφιερωθεί στη δημιουργία του τμήματος αυτού για το δημιουργικό τομέα πριν ξεκινήσει νέο τμήμα μετά το 2025. Τρίτον, να διευκρινιστούν οι προτάσεις όσον αφορά γενικούς και ειδικού στόχους και προς συνάδου με άλλα προγράμματα. Συζητήθηκε, αυτό είναι ένα από τα προβλήματα, ότι δεν εξετάζεται ευρύτερο το Ινστιτούτο αυτό εν συγκρίση με άλλα προγράμματα. Πρέπει να ενταχθεί σε άλλε άλλες δαπάνες για άλλα προγράμματα, όπως ε, για τις ευφυείς πόλεις, και διάφορα άλλα προγράμματα, αυτό είναι ένα κενό, μια έλλειψη που ίσως να μην καλύπτεται με την παρούσα νομοθετική πρόταση, αλλά περιμένουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση του μέσου αυτού. Κάτι πολύ σημαντικό για μένα στη σύνταξη της ήταν η ε, ευθυγράμμιση του πρόγραμμα Horizon Ευρώπη. Πρέπει ο στόχος του EIT να συνδυαστεί με το Horizon Ευρώπη, να δούμε πώς βελτιώνουμε την επιρροή σε περιφερειακό επίπεδο με συμμετοχή περισσότερων φορέων και θα πρέπει να υπάρχουν περιφερειακές στρατηγικές και σχέσεις με στρατηγική για ευφυείς εξειδικεύσεις, ευφυείς ειδικότητε. Ανησυχώ ιδιαίτερα διότι στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων όσον αφορά τα διεθνωτικά ταμεία δεν γίνεται μενία στα διάφορα τμήματα του Ευρωπαϊκού Αυτού Ινστιτούτου Τεχνολογία. Εξετάσαμε όλα τα προγράμματα των κρατών μελών και δεν υπάρχει ούτε μία μενία του EIT. Αυτό είναι παράξενο, είναι πολύ άγνωστο. Από πλευράς Συμβουλίου και από πλευρά ε, διαπραγματευτών και υποπτικών φορέων για τα επιχειρησιακά προγράμματα των κρατών μελών, στα διαθετικά ταμεία θα πρέπει να γίνεται μία μνήα στο EIT. Δεν έχει νόημα να θέλουμε να ανοίξουμε το πλαίσιο του EIT και να το πρικοδοτήσουμε κατάλληλα με χρήματα από τα διαθωτικά ταμεία αν δεν ξέρουν οι διάφορες πλευρές περί τίνος πρόκειται. Πρέπει να αυξηθεί η δυνατότητα καινοτομία της ανώτατη εκπαίδευση, να ενταχθούν αυτοί οι φορεί ε, στα διάφορα τμήματα. Θα πρέπει να έχουμε νέα τμήματα και προτεραιότητε που θα επιλεχθούν ανάλογα με το πόσο σχετική είναι η τομή με τι προτεραιότητε του ορίζοντα Ευρώπη, το, ο πρώτο τομέα που θα ξεκινήσει το 2022 νέος τομέας αφορά τον πολιτισμό και τη δημιουργική βιομηχανία. Για μία ακόμη φορά θέλω να ευχαριστήσω την DGR. Ε, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Ε, ε, είναι κοινή προσπάθεια, λήφθησαν υπόψη οι προτάσεις μας. Ήτρε και Επιτροπή Κολτ συνεργαστήκαμε. Ήμασταν επιτυχεί όσον αφορά αυτό και από την αρχή των συζητήσεων ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε άλλο ήταν πολύ ανοιχτόμυαλος για τι ιδέε που εκφράσαμε. Τώρα θεωρείται κάτι πιθανό αυτό που προτείνουμε. Στην αρχή όμως θυμηθείτε ότι έγινε σκληρή μάχη και δεν υπήρξε καλή συνεννόηση όσον αφορά τη σημασία του δημιουργικού τομέα και κυρίως για το EIT. Πρέπει να προωθούμε την επιχειρηματικότητα, βλέπετε, στο δημιουργικό τομέα και θα πρέπει να το συσχετίσουμε αυτό με τεχνολογία. Και αυτό το τρίγωνο της τεχνολογίας είναι η ιδεώδης πρόθεση για το δημιουργικό τομέα. Στην αρχή ήταν δύσκολα. Στο τέλος ακούγονται έπαινοι βέβαια. Και φαίνεται προφανή η απόφαση. Μη λησμονούμε όμω ότι δόθηκε σκληρή μάχη πάνω σε αυτό και το Κοινοβούλιο έσπροχνε προς αυτή την κατεύθυνση. Και η DGE και άλλες γενικές διευθύνσεις ήταν διστακτικοί. Τελικά υποστηρίχθηκε η πρόταση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η αναδιατύπωση θα κατάλληλα με τον ορίζοντα Ευρώπη για πρώτη φορά στα προγράμματα έρευνας αναφερόμαστε στη δημιουργική βιομηχανία, στο δημιουργικό τομέα και πρέπει να είναι ολοκληρωμένη η προσέγγιση, διότι έχουμε οικονομική μόχλευση έτσι και ουσιαστική πρόθεση του τομέα θα είναι οδυνηρή συζήτηση που θα λάβει χώρα για τα οικονομικά. Πιθανότατα στο δεύτερο εξάμεινο θα γίνει αυτή η κουβέντα, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Το EIT να μην είναι αποδιοπομπέως τράγος στις διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μπάντιν έχει το λόγο. Παρακαλώ. Συγγνώμη, δεν ξέρω γιατί μου δίνετε το λόγο. Για να συνεχίσουμε λοιπόν, η Ντομινίκ δεν είναι στη θέση της και είστε σκιώδες γι' αυτό. Το μόνο σχόλιο είναι ότι ναι, συμφωνώ. Θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί απόλυτα το Ινστιτούτο με το Horizon Europe. Αλλά για να επανέλθω στα θέματα δημιουργικότητας του τμήματος. Θα σας πω ότι εγώ εργάζομαι στα μέσα, στα μίδια και όταν το είδα είπα πω πω μ' αρέσει πάρα πολύ η ενίσχυση των δημιουργικών αυτών κλάδων, αλλά δεν είμαι σίγουρη πως είναι ο κατάλληλος τόπος. Γιατί το EIT θα πρέπει να είναι το MIT της Ευρώπης. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε τις επιχειρήσεις να ε, ε, το κουκουλώσουν, γιατί είναι ένα τεχνολογικό ίδρυμα το οποίο θα πρέπει ουσιαστικά να αφιερωθεί στην τεχνολογία. Αλλά όταν κάνει κανείς όταν το ψάξει κανείς, διαπιστώνει πως η ανάπτυξη των ε, ε, δημιουργικών αυτών επαγγελμάτων που ήταν πετυχημένες σε εμπορικό επίπεδο εκρηκτικά βασίζονται σε τεχνολογικές ε, εξελίξεις. Ε, τα βιντεοπαιχνίδια, τα παρουσιάσεις με ολογράμματα και τρισδιάστατες. Όλα αυτά βρίσκονται στο όριο του να εκτοκτεστούν και δεν θα πρέπει να μείνει πίσω η Ευρώπη δεν θα πρέπει να το επιτρέψουμε και γι' αυτό στηρίζω το να έχουμε ε, τις ε, επιχειρήσεις αυτές, τις βασίζονται στη δημιουργία, να ε, ενταχθούν στο, στα τμήματα αυτά του Ινστιτούτου. Δεν θα είμαι εδώ για να στηρίξω αυτή τη μάχη αργότερα φέτος και δεν ξέρω σε ποιον θα πρέπει να στραφώ. Κρίστιαν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σας παρακαλώ πολύ μην ξεχνιέστε όταν γίνονται οι συζητήσεις αυτές πως αυτοί οι οποίοι ε, θα πούν το ναι ή το όχι ε, είναι αυτοί οι οποίοι ε, ασχολούνται με τα θέματα της δημιουργικής τεχνολογίας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχετε τα στοιχεία στη διάθεσή σας για να τους πείσετε. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Έλερ για την δημιουργική του προσέγγιση. Θέλω να ξεκινήσω με τα πιο σημαντικά στοιχεία για μένα και ίσως και για τη δική μας επιτροπή. Λυπάμαι που επαναλαμβάνομαι, αλλά η δημιουργία αυτού του Ινστιτούτου και των τμήματων ε, για τις καλλιτεχνικούς και δημιουργικούς κλάδους είναι σημαντική για να καταφέρουν τα νέα ταλέντα να βρουν τη θέση τους. Και χαίρομαι που η συγγήτρια το τόνισε, είναι και που ο, εισηγητής, μίλησε ε, για τις προτεραιότητες που δίνει ε, στο σημείο αυτό. Πάντως θα πρέπει να προσπαθήσουν να πετύχουν κάποια οικονομική σταθερότητα. Και επειδή εδώ έχουμε αναπομπή, ε, θα είναι καλύτερα να τονίσουμε πως θα πρέπει το Ινστιτούτο να βοηθήσει αυτά τα τμήματα στη μετάβαση αυτή και αν τα αποτελέσματα που θα παραδώσουν θα είναι ε, ε, ανεπαρκή, θα πρέπει να υπάρχει χώρος και για διορθωτικές κινήσεις. Συμφωνώ πως θα πρέπει να ενταχθούν και τα τμήματα και το Ινστιτούτο και τα σχετικά κέντρα να μπουν ε, μέσα στα διορθωτικά ταμεία για να χρηματοδοτούνται καλύτερα και για τις συντονισμένες εκπαιδευτικές δράσεις να σας πω πως δεν θα πρέπει το Ινστιτούτο μόνο να στηρίζει ε, τα τμήματα αυτά έτσι ώστε να ενταχθούν στην υψηλή αξία παιδεία, αλλά θα πρέπει να δώσουν του κατάλληλου προσανατολισμού, να προσφέρουν συμβουλευτικέ υπηρεσίε, να συμμετέχουν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Και στα πλαίσια αυτά, η απόκτηση των επιχειρηματικών δεξιοτήτων και τη ε, τεχνογνωσία τη καινοτομία είναι σημαντικά. Ε, ο εισηγητή ε, και η συγγήτρια τόνισαν τα στοιχεία αυτά και νομίζω ότι θα καταφέρουμε πολλά περισσότερα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Πρωτού δώσω το λόγο στην Κομισιόν, θέλω εγώ να πω δύο λόγια. Εγώ χαιρετίζω. Α, συγγνώμη. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Uh, just like to make a few... Θέλω να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις που σχετίζονται με τη δουλειά που έκανε η Judith στην προηγούμενη έκθεση και αυτήν. Να μιλήσω δηλαδή για, το, για, τις, για τους κλάδους STEM. Εγώ την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία ε, την πέρασα να σας μιλώ διαρκώς για το STEM και όχι για το STEM. Και είμαι πραγματικά πολύ περήφανη που πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση μιλά για STEM Και σας καλώ να συνεχίσετε αυτήν την κουβέντα. Δεν μπορούμε να χάσουμε το α τις ανθρωπιστικές σπουδέ δηλαδή, χρειάστηκαν χρόνια για να αναγνωρίσουν οι άνθρωποι ότι οι ανθρωπιστικές σπουδέ είναι ύψης της σημασίας για την κοινότητα STEM και οι διαφορές ανάμεσα, στην, στην, οι διαφορές ανάμεσα στους ε, δημιουργικούς κλάδους και τους επιστημονικούς κλάδους είναι τελείως τεχνητοί. Χρειάζεται και οι ίδιοι οι επιστήμονες να είναι δημιουργικοί και το αντίθετο συμβαίνει. Οι δημιουργικοί άνθρωποι του πολιτισμού χρησιμοποιούν μαθηματικά, χρησιμοποιούν φυσικούς νόμους, οι αρχιτέκτονες ε, χειρίζονται τον χώρο και τον διαμορφών, οπότε οι ανθρωπιστικές και οι θετικές επιστήμες είναι ένα ενιαίο σύνολο. Ο διαχωρισμός τους είναι τεχνητός πάντοτε. Γι' αυτό και θέλω να σας ε, επιστήσω την προσοχή και στην ε, οργάνωση Insignia που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά έχουν ε, συντάξει και μελέτες και ε, ε, κάποια έγγραφα με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Το Νέστερ από το Ηνωμένο Βασίλειο που επίσης είναι ένας, μια οργάνωση ηγέτιδα στο Ηνωμένο Βασίλειο που ασχολείται και δραστηριοποιείται στον τομέα του πολιτισμού και των επιστημών. Επίσης υπάρχει οργάνωση χίλιες και μία καινοτομίες που προσπαθεί να αναδείξει τον ιστορικό ρόλο και την ιστορική σχέση που είχε ο Ισλαμικός κόσμος, ο μουσουλμανικός κόσμος ε, στον τομέα της επιστήμης, της αρχιτεκτονικής, του πολιτισμού, της ιατρικής, της υγείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και στο υπάρχον, στην υπάρχουσα ατμόσφαιρα που έχει γίνει πολύ Ισλαμοφοβική, ε, ιδίως στη δική μου χώρα και ξέρω ότι και σε ολόκληρη την Ευρώπη ε, υπάρχει αυτό το πρόβλημα άνθρωποι να μην αναγνωρίζουν αυτήν την ποικιλόμορφη κληρονομιά που έχει η Ευρώπη. Οπότε ε, εγώ έχω προσκαλέσει και τον διευθυντή αυτής της οργάνωσης, τον, τον είχα προσκαλέσει στην προηγούμενη θητεία αυτής της οργάνωσης, της ε, οργάνωσης χίλιες και μία ε, ανακαλύψεις και ώστε να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε αυτή την άρνηση της συμβολής του μουσουλμανικού κόσμου στον πολιτισμό και τις επιστήμες στην Ευρώπη. Οπότε θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει κανείς να εξετάζει το ζήτημα αυτό ολιστικά και τις ανθρωπιστικές σπουδές λοιπόν και τις θετικές. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλω και εγώ τώρα να τοποθετηθώ, να ευχαριστήσω τον κύριο Έλερ που κατάφερε να φέρει ε, στο επίκεντρο της προσοχής και τους ε, πολίτες, τους δημιουργικούς τομείς. Διότι, διότι δυστυχώς στο παρελθόν ε, είναι, είναι γνωστό ότι ο πολιτισμός, η δημιουργική κλάδη συνέβαλαν σημαντικότατα και στην τεχνολογική εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Στην, στην τηλεόραση, για παράδειγμα, στα παιχνίδια, όλα αυτά ε, κινητοποιήθηκαν και τους δόθηκε ζωή από ανθρώπους δημιουργικούς. Ε, δεν θα είχαν γίνει αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις αν δεν είχε προηγηθεί η ιδέα και η δουλειά των ανθρώπων που ασχολούνται με τον πολιτισμό. Είναι πραγματικά ε, σχεδόν τρομακτικό πόσο η τεχνητή νομιμοσύνη έχει εισχωρήσει πλέον και στις δημιουργικούς, στους κλάδους. Οπότε πράγματι είναι σημαντικό να δοθεί ειδική, εξειδικευμένη προσοχή για το πώς μπορεί να συγχωνευτεί ο δημιουργικός κλάδος, η δημιουργική κλάδη εν γέννη με, την, με τους τεχνολογικούς κλάδους. Γι' αυτό και θα πρέπει να εξετάσουμε το πράγμα ολιστικά. Όχι να δημιουργήσουμε ένα κέντρο, ένα τμήμα για τον, για τον πολιτισμό και τη δημιουργία, αλλά ένα ενιαίο κέντρο το οποίο θα μπορεί να συγχωνεύει και να συνδυάζει την τεχνολογία και τον πολιτισμό, ώστε με τη σειρά τους αυτά τα κέντρα στη συνέχεια να μπορούν να αναπτύσσουν ε, έργα και project τεχνολογικό-πολιτιστικά Γι' αυτό και αυτό που είπε η Τζούλι Ward είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για STEM, για θετικές επιστήμες, αλλά για STEAM μαζί με τις ανθρωπιστικές επιστήμες δηλαδή. Ακριβώς για να συνδυάζεται πάντοτε η τεχνολογική εξέλιξη με τη δημιουργία, με τον πολιτισμό, να υπάρξει δηλαδή αυτή η οριζόντια σκέψη, αν θέλετε, η οποία θα συνδυάζει ε, τους διάφορους κλάδους ανθρώπινης δραστηριότητας και του ανθρώπινου πολιτισμού. Το βλέπει κανείς και στα πανεπιστήμια που προσφέρουν τμήματα και θετικά και ανθρωπιστικά. Έχουν πάντοτε τα πανεπιστήμια αυτά, αυτά τα ικανομαϊκά ιδρύματα, μια πολύ διαφορετική προσέγγιση απέναντι και στάση απέναντι στα πράγματα, στις κοινωνικές υποθέσεις για παράδειγμα, αν τα συγκρίνει κανείς με ιδρύματα που εξειδικεύονται μόνο στην τεχνολογία. Αυτά από μένα. Να δώσω ξανά το λόγο στην ε, Κομισιόν και στη συνέχεια θα σας δώσω, ε, κυρία εισηγήτρια, τον λόγο ξανά. Ευχαριστώ, λέει η εκπρόσωπο. της Κομισιόν. Σας ευχαριστούμε πραγματικά και χαιρετίζουμε αυτήν την εξαιρετικά θετική ε, στάση σας απέναντι στο CCI KIC. Από εμά είναι ξεκάθαρο ότι το α στο STEAM θα διατηρηθεί και ότι οι δημιουργικοί κλάδοι βεβαίως και θα ε, έχουν την δέουσα προσοχή, την προσοχή που τους ε, αρμόζει και θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να μπορέσει να υπάρξει μια καλή συνεργασία. Επίσης χαιρετίζουμε τις θετικές σας απαντήσεις όσον αφορά την αύξηση των ε, ικανοτήτων, των ερευνητικών ικανοτήτων των ε, ανώτατων ιδρυμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αυτό είναι ένας στόχος τον οποίο θα επιδιώξουμε και εμείς με όλες μας τις δυνάμεις. Επίσης, είμαστε ε, πολύ θετικοί απέναντι σε αυτήν την ε, πρόταση ανοίγματο των ΣΚΙΚΣ. Ε, είμαστε και εμείς υπέρ της υψηλότερης διαφάνειας. Είναι ένας στόχος που τον έχουμε βάλει και εμείς στην Κομισιόν μέσω του μηχανισμού ερευνητικής και έρευνας και κοινοτομίας. Όσον αφορά την, τον, την ευθυγράμμιση με τον ορίζοντα Ευρώπη, δεν διαφωνούμε, όμως πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο κανονισμός EIT θα συνεχίζει να βασίζεται σε αρχές, ενώ όλες οι λεπτομέρειες ε, θα παραμένουν στο SIA. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια καινούρια ε, ισορροπία για το πώς ακριβώς θα μπορέσουν να ενταχθούν στον κανονισμό αυτά τα καινούρια τμήματα. Προσπαθούμε από πλευράς Κομισιόν να ε, γίνουν όλα αυτά ουδέτερα από άποψη χρόνου, γι' αυτό όλα θα πάνε στο SIA. Έχουμε και μία αύξηση του προϋπολογισμού που προτείνεται τη τάξη του 4%. Το σημειώνουμε. Εμείς έχουμε υποβάλει συγκεκριμένη πρόταση προϋπολογισμού, αλλά είναι κάτι το οποίο είχαμε ήδη συμπεριλάβει με ένα 25% αύξηση σε σχέση με το Horizon 2020. Καταλαβαίνουμε όμως και κατανοούμε πως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να κάνει μία αύξηση γύρω στο 4%. Πάντω, γενικά πρέπει να σα πω πω στηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό την πρότασή σα. Ωραία, ευχαριστώ. Οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο. Όχι. Ναι. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 27 Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι. Και επίσης η ψηφοφορία για αυτό το θέμα θα γίνει στις 17 Φεβρουαρίου. Όχι, συγγνώμη, πάλι μπερδεύτηκα. 27 Απριλίου. Αλλά μπορεί να γίνει ψηφοφορία και στις 17 Μαρτίου εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού. Οπότε θα δούμε, θα δούμε. Δεν υπάρχει πάντω πρόβλημα, χρόνο υπάρχει, θα δούμε πώ θα διαμορφωθεί η ημερήσια διάταξη. Πάντω προθεσμία για τροπολογίε 27 Ιανουαρίου. Σημείο 8. Εξέταση γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμενο για το Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών, Απασχόληση και Κοινωνικέ Πτυχέ στην ετήσια επισκόπηση τη ανάπτυξη για το 2020. Θα θυμάστε ότι οι συντονιστέ είχαν αποφασίσει η Επιτροπή μας να συντάξει γνωμοδότηση για αυτήν την ε, ε, έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας της Επιτροπής Απασχόλησης πριν από την Σύνοδο Κορυφή ε, την Εαρνή του 2020 θέλουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά με την έκθεση. Αυτό είναι και ο στόχος μας. Βάση αυτή τη ε, έκθεση είναι η ανακοίνωση Κομισιόν για την απασχόληση και κοινωνικέ πτυχέ στην ετήσια επισκόπηση τη ανάπτυξη για το 2020. Και εδώ ε, πρόκειται για έναν, μια έκθεση εργασίας για την απασχόληση. Εκεί σε αυτή την έκθεση ε, σκιαγραφούνται τα βασικότερα στοιχεία σχετικά με την απασχόληση στα κράτη-μέλη. Περιλαμβάνει και κάποιες προτάσεις για τη βελτίωση των ικανοτήτων όπως είναι η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η βελτίωση του μορφωτικού επίπεδου και ε, ο συνδυασμός αυτών με την ε, απασχόληση. Λόγω του χρονοδιαγράμματος της Επιτροπής Απασχόλησης, η γνωμοδότηση και η συζήτηση μπορεί να γίνει μόνο στα αγγλικά. Η ισοφορία στην ΕΜΠΛ θα γίνει στις 20 Φεβρουαρίου, οπότε η γνωμοδότησή μας θα πρέπει να έχει εγκριθεί έως τις 19 Φεβρουαρίου, δηλαδή στην επόμενη συνεδρία τη Επιτροπή μα, ώστε να μπορέσει να τη λάβει υπόψη τη Επιτροπή Απασχόληση. Το 2019 ε, το κάθε κράτο μέλος έλαβε συγκεκριμένες συστάσεις για την εκπαίδευση, ανάπτυξη ικανοτήτων, διαβίου μάθηση, καθώς και έρευνα και κοινοτομία για όλους αυτούς τους τομείς. Το σχέδιο που έχετε λάβει, που είναι όπως είπα στα αγγλικά, γιατί πρέπει δυστυχώς να ε, ε, προχωρήσουμε γρήγορα, ε, γι' αυτό και θα αρχίσω να θα γυρίσω στα αγγλικά. Λοιπόν, μετά την ε, αποστολή σε εσά του σχεδίου, τα στοιχεία είναι τα εξή. Καλούμε την ε, Ευρωπαϊκή Κομισιόν να και τα ευρωπαϊκά κράτη να προσαρμοστούν εν ώψη των προκλήσεων που θέτουν η ψηφιοποίηση και η τεχνητή νομιμοσύνη αναδεικνύουμε ότι οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες είναι ε, παράγοντας ε, κακών οικονομικών αποτελεσμάτων, οπότε πρέπει να ε, επιμείνουμε στην ποιοτική εκπαίδευση. Χρειάζεται η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, όχι μόνο ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά χρειαζόμαστε μια ευρύτερη προσέγγιση για τον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευση. Όχι για να εξισωθούν τα πάντα, αλλά τουλάχιστον να γίνουν συγκρίσιμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι, είναι σημαντικό να το αποκτήσουμε αυτό ως αποτέλεσμα, να υπάρχουν δηλαδή συγκρίσιμα αποτελέσματα και ε, εκπαιδευτικές δομές. Πώς να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες. Χρειάζεται να ε, δοθεί έμφαση στην προσχολική αγωγή, ε, ιδίως για εκείνα τα παιδιά που έχουν ε, λιγότερες ευκαιρίες λόγω του κοινωνικού τους, της κοινωνικής τους καταγωγής προέλευσης είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει προσχολική αγωγή ώστε να έχουν τα παιδιά αυτά τη δυνατότητα και την ευκαιρία να εισέλθουν με τον κατάλληλο τρόπο στο εκπαιδευτικό σύστημα. Για να ε, αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων, τονίζουμε τη σημασία που έχει η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, ώστε να δοθούν κίνητρα και να ενθαρρυνθούν οι νέοι άνθρωποι να ανοίξουν τις δικές τους επιχειρήσεις, δηλαδή όχι μόνο το κλασικό αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων, αλλά ε, να δημιουργηθούν και δεξιότητες και εργαλεία ε, δημιουργικότητας ώστε ένα παιδί να μπορεί να γνωρίζει πώς μπορεί να κάνει μια επιχείρηση όταν δεν μπορεί για παράδειγμα να βρει μια δουλειά. Τα κράτη-μέλη πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων για να αντιμετωπιστεί το χάσμα, η έλλειψη δεξιοτήτων. Εγώ δεν θέλω τα σχολεία βεβαίω να αντικατοπτρίζουν μόνο τι ανάγκε των επιχειρήσεων, όμω αν δεν το κάνουν και καθόλου, επίση δεν είναι καλό. Οπότε χρειαζόμαστε μια ισορροπία. Για να, υπάρχουν, για να υπάρχει το γενικό σύνολο δεξιοτήτων και γνώσεων, το οποίο θα παρέχεται στα παιδιά μέσω των σχολικών συστημάτων των εκπαιδευτικών συστημάτων, αλλά με κάποιον τρόπο όλα αυτά να αντιστοιχίζονται και στις ανάγκες της αγοράς. Αποτελεσματικότητα της επαγγελματική εκπαίδευσης. Επίσης, αυτό αφορά κυρίως τους, τις μη προνομιούχες ομάδες του πληθυσμού, μετανάστες και αποτελεί και έναν πυλώνα για την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και πρέπει επίσης να δώσουμε προσοχή ε, στους ε, ανθρώπους που εγκαταλείπουν πρόωρα τα σχολεία, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι και αυτό ένας παράγοντας που ενισχύει την ανεργία σε πολλές χώρες. Υπάρχουν χώρες όπου υπάρχουν πάνω από 10% των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο πριν από την ώρα τους. Είναι και αυτό ένα τομέας στον οποίο πρέπει να εργαστούμε. Αυτό ήταν και ένα θέμα που είχε απασχολήσει και την ατζέντα της Λισαβόνας είναι λοιπόν μια δουλειά η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αλλά παρά το γεγονός αυτό ότι, ήδη, ότι εδώ και χρόνια δίνεται έμφαση σε αυτό, υπάρχει ακόμη πάρα πάρα πολλή δουλειά που πρέπει να γίνει για να μπορέσει να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτά τα θέματα νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρονται και στην έκθεση, ε, προφανώς μέσω της γνωμοδότησης που έχουμε τη δυνατότητα να συντάξουμε, είμαστε κάπως περί περιορισμένη, όμως ε, προσβλέπω στο να λάβουμε κάποιες ε, καλές προσθήκες, θετικές προσθήκες και από την δική σας πλευρά, καθοδόν προς την ε, σύνταξη και την έγκριση αυτής της γνωμοδότησης από την Επιτροπή Πολιτισμού. Η Πέτρα Καμερέβερτ από τους Σοσιαλιστές έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να, σας, ζητήσω συγγνώμη εκ μέρους της κυρίας η οποία παρουσιάζει έκθεσή τη στην Επιτροπή προπολογισμού. Γι' αυτό και δεν είναι εδώ. Όμω μου έδωσε κάποιε παρατηρήσει τι οποίε θέλω εδώ να σας ε, ε, παρουσιάσω. Ε, Καταρχά, εκ μέρου τη κύρια Βόλτα, θέλω να σα να σας ευχαριστήσω για την εξαιρετική σα γνωμοδότηση. Νομίζω ότι αναδεικνύονται οι βασικέ προκλήσει που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στον τομέα τη εκπαίδευση και η κυρία Βόλτα. Ε, θέλει να δοθεί ιδιαίτερη έμβαση στην κοινωνική ένταξη όλων των ε, πολιτών. Η κοινωνική ένταξη, η κοινωνική συνοχή αποτελούν στοιχεία που θα εξασφαλίσουν την προετοιμασία της κοινωνίας μας ενώ προκλήσεων όπως είναι η ψηφοποίηση και τη τεχνολογική νοημοσύνη. Στη βάση όλων αυτών η Λάρα Βόλτας θα ήθελε να αντικατοπτρίζονται δύο σημεία στις τροπολογίες. Πρώτον, πώς θα ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να κάνουν επαρκείς επενδύσεις στην εκπαίδευση και πόσο απαραίτητο, ε, θα το δούμε και το απόγευμα σήμερα αυτό, όταν θα παρουσιαστεί η τελευταία έκθεση πίζα, πόσο σημαντικό ε, είναι το γεγονός και πόσο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι όλα τα, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη ε, βρίσκονται πλέον σε μια φθήνουσα πορεία όσον αφορά τα εκπαιδευτικά του αποτελέσματα. Είναι αυτό μια μεγάλη πρόκληση. Οπότε πρέπει και ω Κοινοβούλιο να ασκήσουμε μεγάλη πίεση στα κράτη-μέλη για να ενισχυθούν οι επενδύσει. Και δεύτερον, πώ. Το ερώτημα, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η εκπαίδευση και η επαγγελματική εκπαίδευση θα έχει τον, ε, τη θέση που δικαιωματικά της ανήκει και στην Πράσινη Συμφωνία, η οποία αποτελεί πλέον το μεγάλο θέμα συζήτησης, Πώς θα γνωρίζουν οι άνθρωποι ότι με τις ε, δεξιότητες τους, τις γνώσεις τους θα μπορέσουν να συμβάλλουν σε αυτούς τους πράσινους στόχους και πώς, μπορούμε, πώς θα μπορέσουμε να ε, ε, ενισχύσουμε και καινοτόμες πράσινες λύσεις για το μέλλον. Η Λάρα Βόλτες, ε, σας ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία, προσβλέπει την περαιτέρω συνεργασία μαζί σας και με τους υπόλοιπους σκιώδεις. Αυτά. Ο η Ντάτσα Μαλβάρντε έχει το λόγο. Ε, ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευπρόσδεκτη έκθεση. Επενώ τη συνοπτική της μορφή. Ποιοτική παιδεία και κατάρτιση είναι πρωτής της σημασίας εν τη προετοιμασία για την ψηφιοποίηση και τον αυτοματισμό. Παρομοίως, η έκθεση σωστώς εντοπίζει σειρά άλλων συναφών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η αγορά εργασία. Δεξιότητε που δεν ταιριάζουν στι απαιτήσει, ανεπαρκή επίπεδα εκπαιδεύσεω, πολύ συχνά αυτό οφείλεται σε κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο και έλλειψη συνεργασία μεταξύ ανώτατη παιδεία και επιχειρήσεων. Και συμφωνώ απόλυτα χρειάζονται καθηγητές και δάσκαλοι με περισσότερα κίνητρα Χρειάζεται ισορροπία των φύλων, να έχουμε περισσότερους άντρες δασκάλους σε κάποια κράτη-μέλη, διότι υποεκπροσωπούνται σε πολλά κράτη-μέλη οι άντρες καθηγητές και δάσκαλοι. Για την απασχόληση και την κατάρτιση και παιδεία υπάρχουν διαφορές μεταξύ κρατών μελών και το σημαντικότερο και εντό των κρατών μελών υπάρχουν διαφορές. Η εκπαιδεία και επιτεύγματα και στατιστικές για την απασχόληση δίνουν ανησυχητικά στοιχεία αν δούμε τι γίνεται με απόμακρες περιοχές σε σύγκριση με τις πόλεις. Αναλύοντας και τα επίπεδα ανεργίας, βλέπουμε ότι η ανεργία των νέων παραμένει πολύ υψηλή. Η συζήτηση συνήθως αφορά το θέμα δουλειάς υποαπασχόλησης και ενεργίας και επισφαλούς απασχόλησης. Οι άλλοι τομείς επισφαλούς απασχόλησης θα πρέπει να εξετάζονται εκεί που ε, και αυτή η γκρίζα ζώνη εκείνων που μας οδηγούν στη, στην πόλη και μας πηγαίνουν σε διάφορες διαδρομές και μας παραδίδουν τρόφιμα ε, και έχουν επισφαλή μορφή εργασίας, αυτή θα επέλεγα μια πιο ασφαλή και μόνιμη εργασία αν είχαν την ε, δυνατότητα να διαλέξουν. Όσον αφορά το επικείμενο κείμενο αυτοματισμού, αυτοματοποίησης, υπάρχουν διάφορες ομάδες εκτός από τις μειονεκτούσες ομάδες που πρέπει να εκπαιδευτούν Χρειάζεται αναβάθμιση δεξιοτήτων και αλλαγή δεξιοτήτων, διότι αλλάζουν ε, τα είδη της εργασίας και εκείνοι που φτάνουν στο επίπεδο συνταξιοδότησης και εκείνοι που ε, έχουν ανεπαρκή εκπαίδευση πρέπει να προσαρμοστούν. Χρειάζεται πάλι ισότητα των φύλων. Συζητώντας τις απώλειες θέσεων εργασίας που επίκειται, ε, στη βιομηχανία οι άντρες έχουν περισσότερες θέσεις απασχόληση και αυτέ προσέχονται περισσότερο. Εκεί που ασχολούνται περισσότερο, απασχολούνται οι γυναίκες, οι θέσεις αυτές δεν συζητώνται πολύ συχνά για τις δεξιότητες. Δεν πρέπει να αναφέρουμε μόνο τις ψηφιακές και παλαιότερες δεξιότητες. Κριτική σκέψη, γνώση για τα διάφορα μέσα, δυνατότητα να αργάζεσαι σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον, χρειάζεται και συναισθηματική ευφυΐα. Αν τα προσθέσουμε τα στοιχεία αυτά, η έκθεση γίνεται πληρέστερη. Και προσβλέπω και στην ε, επικοδομητική εργασία που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μόνικα Σεμέντο, νέο μέλος της Ρινιού. Και θα αναλάβει επίσης και τη θέση σκιώδου για το Ρινιού. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά. Είμαι η Μόνικα ε, Ζεμέντο, νέο μέλος ε, εκ μέρους του Renew και είμαι εδώ στην Επιτροπή Πολιτισμού από λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Χαίρομαι πολύ για όλα τα θέματα που εξετάζει. Μόλις χθες ε, ορίστηκα ως σκιώδης για αυτήν την γνωμοδότηση και προσπάθησα να εξοικειωθώ λίγο με το θέμα, δεν είχα όμως πολύ χρόνο να σας πω, οπότε δεν έχω και κάποιες συγκεκριμένε τροπολογίες, όμως το επόμενο διάστημα θα το κάνω και αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ που αναφέρατε τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης. Είναι κάτι που το υποστηρίζω και εγώ πλήρως. Για να υπάρξει έτσι μια προσέγγιση Θέλω όμως να τονίσω και θα το κάνω και στις ε, τροπολογίες μου ότι η αμοιβαία αναγνώριση δεξιοτήτων και πτυχίων είναι ένα στοιχείο κρίσιμο για την ε, ενίσχυση της ε, κινητικότητας στην Ευρώπη. Θα είναι αυτός ένας τομέας στον οποίο θα εστιαστώ ιδιαιτέρως, αλλά θα τα πούμε και στις τροπολογίες. Για τους πράσινους δεν έχουμε κάποιον λέει πρόεδρος, οπότε να δώσω το λόγο στους ε, υπόλοιπους συναδέλφους. Αν θέλει κάποιος να τοποθετηθεί, να παρέμβει, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για... Ευχαριστώ πολύ για πολύ ενδιαφέροντες ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις που ακούσαμε. Όμως, η στενή σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και ε, εκπαίδευσης ε, με ανησυχεί. Γιατί πολλές φορές απευθύνονται στους μαθητές σας σχολεία ε, με διδασκαλία που ουσιαστικά προσεγγίζει τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Και δεν μπορεί κανείς να σπουδάσει ελεύθερα όταν το μόνο που τον ανησυχεί είναι η θέση που θα καταλάβει στην αγορά εργασίας. Και παρόλο που σε μια προηγούμενη συζήτηση μιλούσαμε για τις βιομηχανίες του θεάματος και τις δημιουργικές βιομηχανίες, θεωρώ πως παρόλα αυτά θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε και να μην... ε, ε επιτρέψουμε να κατηγορηθούν όσοι ασκούν τέχνες ως αχρηστοί ε, και ανειδίκευτοι. Και ξέρετε πως πολλές φορές από τη σχολική ύλη, από τις εξετάσεις, αφαιρούνται τα μαθήματα τέχνης γιατί δεν θα βοηθηθούν όσοι τα ακολουθούν να βρουν μετά δουλειά. Αυτό είναι ανησυχητικό για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και πάντα βέβαια όταν ζητάμε από τα σχολεία ε, να κατευθύνει τους ε, μαθητές να κατηγορηθούμε πως ζητάμε να προπαγανδίσουν. Γιατί όταν τους ζητάμε να μιλήσουν για δημοκρατία, ποια δημοκρατία θα πρέπει να προωθήσουν. Και αυτό το ζητάμε σε όλη την Ευρώπη με την ίδια ένταση. Το λέω γιατί είναι θέματα εξαιρετικά λεπτά και δεν θα ήθελα κανείς να ε, προωθεί συγκεκριμένη πολιτική σχολή σκέψης στα σχολεία. Γι' αυτό κάνω αυτή την παρατήρηση. Νομίζω πως στην ε, αναφορά, στην έκθεση αυτή δεν υπάρχει καμία ε, υποψία προπαγάνδα στην οποία εμείς ε, θα παροτρύνουμε στα σχολεία ή που θα επηρεάζουμε τα σχολεία μέσω επιχειρήσεων. Τα σχολεία θα πρέπει να είναι αυτόνομα και θα είναι ένας πύργος γνώσης που όμως δεν θα πρέπει να είναι παντελώς αποκλεισμένοι από τον κόσμο γύρω τους Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι με τον οποίο μπορούμε να προωθήσουμε τη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Οι βασικές αρχές πάντως της δημοκρατίας θα πρέπει να εξηγούνται και να αποτελούν ε, ε, να πόσπαστα στοιχεία των όσων διδάσκουμε σε ευρωπαϊκά σχολεία με τη γνώση, με τις ευρωπαϊκές αξίες τις οποίες όλοι συμμεριζόμαστε και θα πρέπει τα σχολεία να στέλνουν το μήνυμα αυτό με το σωστό τρόπο και χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική ε, παρέμβαση. Είπα πως είναι πολύ σημαντικό τα σχολεία να αντιμετωπίζουν και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, να προσφέρουν τις δεξιότητες που χρειάζονται, να λαμβάνονται αυτά υπόψη. Αλλά όχι μόνο αυτό, θα πρέπει να προσφέρουν και τις γενικές γνώσεις με, μια, με ένα λογικό μείγμα. Δεν είναι κακό τα σχολεία να έχουν επαφές με τις επιχειρήσεις. Έχουμε πολύ θετικές εμπειρίες από αυτό στη Γερμανία. Για τους νέους, οι οποίοι δυσκολεύονται να περάσουν μετά από το σχολείο στη δουλειά, στον κόσμο της εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να τους προσφέρουμε επαγγελματική κατάρτιση έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν και ε, στα μαθητείας και να έχουν τις δεξιότητες που χρειάζονται γιατί τα σχολεία μπορεί να συνεισφέρουν με άλλες δεξιότητες και γνώσεις αλλά τα παιδιά αυτά κάποια στιγμή θα πρέπει να βρουν και μια δουλειά. Δεν νομίζω ότι είναι λανθασμένη λοιπόν τακτική να υπάρχουν τέτοιου είδους επαφές μεταξύ επιχειρηματικού κόσμου και σχολείων, αλλά με έναν τρόπο που ε, δεν θα επηρεάζει ε, τα σχολεία, δεν θα κάνει επιλογές για τα σχολεία, αυτή η ομή παρέμβαση ε, δεν επιτρέπεται, αλλά θα πρέπει τα σχολεία να έχουν συγκεκριμένου κανόνε. Τα κράτη-μέλη έχουν τελείω διαφορετικού τρόπου όπου αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά, όπου κρίνεται απαραίτητο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για εμά εδώ να μπορέσουμε για τους μαθητές οι οποίοι έχουν λιγότερες ευκαιρίες στη ζωή να ε, αποκτήσουν μια μεγαλύτερη ευκαιρία διείσδυσης στην αγορά εργασίας και με τον τρόπο αυτό να καταπολεμήσουμε και να αποφύγουμε την ανεργία των νέων. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία... Ε, μιλήσαμε. Ε, Κλέρ, δεν συμφωνούμε σε πολλά, αλλά στον περιορισμό της σχολικής ύλη θα συμφωνήσω. Αυτό είναι ε, μεγάλο πλήγμα για τις μέλουσες γενιές και τη δυνατότητα που θα έχουν να είναι ανεξάρτητες, να είναι αυτόνομες, να κάνουν ερωτήσεις, να λύνουν προβλήματα, να συνεργάζονται. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το σημείο αυτό. Ήμουν διευθύντρια σχολείου και έχω εμπειρία από το τι συμβαίνει να δουλεύεις σε ένα σχολείο και να προσπαθείς να δεις ευρύτερα τη λειτουργία του σχολείου αυτού και το είδος των σχέσεων που χρειάζονται να ε, δημιουργηθούν με την ευρύτερη κοινωνία. Είναι σημαντικό τα σχολεία να έχουν αυτή την ευρεία προσέγγιση που είναι ανοιχτή σε όλους, που κάνουν κινήσεις εξωστρέφειας και όταν μιλάμε για επιχειρήσεις, εδώ έχουμε και τις κοινωνικές επιχειρήσεις. Δεν έχουμε μόνο τις κερδοφόρες ή τις μεγάλες επιχειρήσεις. Για παράδειγμα, εγώ ανησυχούσα ιδιαίτερα όταν μεγάλες επιχειρήσεις όπως πετρελαϊκές εταιρείε ή στρατιωτικές ε, δομές προσπαθούν να σε προσεγγίσουν και δεν έχεις κάποια μέθοδο εξορροπήσης. Οπότε θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το ευρύτερο φάσμα του, που καλύπτουμε υπό τον όρο επιχειρήσει ή επιχειρηματικό κόσμο. Και για κάποιον σαν για μένα που έχει μιλήσει με τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στην πιο δύσκολη θέση, που έχουν ξεφύγει από κάθε δίκτυο ασφαλεία το οποίο έχουμε στήσει εμεί, που αποκλείονται από οποιοδήποτε είδους δράση και όπου δεν είχαν καμία ε, αίσθηση ελπίδα για το μέλλον, πρέπει να σας πω πως όντως τα ευρωπαϊκά projects τα οποία, ε, με τα οποία εγώ συνεργάστηκα δεν προπαγάνδισαν καθόλου. Αντίθετα, πρόσφεραν στους νέους ανθρώπους με ε, την απαραίτητη αίσθηση αξιοπρέπειας, ε, γνώσης, δεξιότητας και πραγματικά την αίσθηση της δικής τους τη συνέστηση της δικής τους αξίας και αυτό και παιδιά με αυτισμό, με ε, δυσκολίες μάθησης ε, μπορώ να σας δώσω παραδείγματα ε, με το Headway, το θέατρο Headway στην περιοχή Northumberland όπου κάναμε κάποια project που χρηματοδοτήθηκαν από το Erasmus Plus και τα παιδιά αυτά αισθάνθηκαν αξιοπρέπεια, την οποία την έλαβα μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων και όχι μέσω των όσων τους προσέφερε ή δεν του προσέφερε ποτέ η Βρετανική κυβέρνηση. Στο Stockport, στη δική μου εκλογική περιφέρεια, παιδιά με αυτισμό, Erasmus Plus, εγώ δεν τα συνάντησα στο Stockport, συνάντησα εδώ στι Βρυξέλλε όταν ήρθαν με άλλους αυτιστικούς από την υπόλοιπη Ευρώπη και όταν πήγαν να τους δώσουν το σχολείο τους στο Στόκπορτ αργότερα είχαν προγράμματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, έμπαιναν στην αγορά εργασίας μέσω άσκησης, είχαν στήσει κηλικία ε, και καφετέριες στη δική τους κοινότητα. Αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή προπαγάνδα, αυτό είναι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και οι αξίες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας που ε, ε, ασπάζεται και η επόμενη γενιά. Και με είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι που άνθρωποι σαν εσάς ε, αφαιρούν τις δυνατότητες αυτές από τα παιδιά που είναι αποκλεισμένα στη χώρα μας. Κοιτάξτε, δεν θα κάνουμε Βρετανο-Βρετανική συζήτηση εδώ. Πρέπει να συζητήσουμε το θέμα, το φάκελο και όχι οι βρετανικά πολιτικά θέματα. Κυρία Φόξ, παρακαλώ στα πλαίσια τη ε, έκθεση. Συμφωνώ και αυτό έκανα όταν μίλησα. Ε, για να είμαστε δίκαιοι. Δεν θα απαντήσω σε αυτό το σχόλιο. Ήθελα να διευκρινίσω το θέμα τη δημοκρατία. Κατανοώ ότι είναι σημαντικό να βάλετε υπόψη η δημοκρατία και να κατανοούν τα νέα παιδιά δημοκρατία. Εγώ δεν έκανα κάποια, κάποιο επιθετικό σχόλιο. Εγώ αναφερόμουν στο ότι με τη δασκαλία της δημοκρατίας προβάλλονται διάφορα επιχειρήματα. Μπορούμε τουλάχιστον να δεχθούμε ότι υπάρχουν πολλές απόψεις για τη δημοκρατία και πώς εφαρμόζεται. Για κάποιους π.χ. το Brexit είναι δημοκρατικό, για άλλους όχι. Τι θέλω να πω, ότι αυτό που φαίνεται σαν κάτι αυλαβές να πει κανείς, ε, το θέμα της πολιτικής αγωγής στα σχολεία, σε διάφορες χώρες η δασκαλία εκεί μπορεί να μιλήσει διαφορετικά. Λέω ότι πολύ συχνά η παιδεία στα σχολεία. Και ήμουν δασκάλα πολλά χρόνια. Και εργαζόμουν με τα πιο στερημένα παιδιά, τους μαθητές. Αυτό είναι το ιστορικό μου. Λοιπόν, λέω ότι δούλευα στην παιδεία και έβλεπα πώς οι διάφορες κυβερνήσεις προσπαθούν να χρησιμοποιούν τα σχολεία σαν τρόπο να προωθούν τα δικά τους πολιτικά προγράμματα. Και έλεγα ότι αυτό πρέπει να το προσέχουμε. Επειδή όλοι οι άλλοι το έκαναν, ήθελα να πω ότι παρόλο που φεύγω και χαίρομαι που φεύγω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Κοινοβούλιο αυτό, αντιμετωπίστηκα πάντα με σεβασμό από τους συναδέλφους ευρωβουλευτές, λιγότερα του Βρετανού από του Ευρωπαίου πρέπει να το πω αυτό, και είστε ευπρόσδεκτοι σε όλε τι επιτροπέ που είμαι. Και ήμουν πάρα πολύ ευπρόσδεκτη στι επιτροπέ που μετήχα. Ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Είμαι υπέρ τη Ευρώπη. Θα έχω σχέσει με την Ευρώπη αφού αποχωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι κατά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά είμαι φιλοευρωπαία και θεωρώ ότι είμαι Ευρωπαία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα απόλαυσα, απόλαυσα τη θητεία μου εδώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Φόξ. Ο κ. Μοχάμετ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια στην αρχή της συνεδριάσεως σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα, όπως ανέφερα Ανέφερα και οι συνάδελφοι, εξακολουθώ να εργάζομαι με νέου και θα συνεχίσω όταν επιστρέψω στο Ηνωμένο Βασίλειο στο τέλο τη εβδομάδας με σε άτυπε μορφέ. Και σκοπός μας εδώ είναι να δούμε τι γίνεται σε διάφορες χώρες. Κάποιοι νέοι φεύγουν από, από το δίκτυο της επίσημης παιδείας και μπαίνουν στην άτυπη παιδεία που τους μαζεύει. Και καμιά φορά είναι πολύ ευάλωτοι. Όποια προγράμματα και αν έχουμε, σας απευθύνω έκκληση να θυμόσαστε ότι υπάρχει παράθυρο και για την άτυπη εκπαίδευση. Τα θέματα της ηθαγένειας, της πολιτικής αγωγής θα πρέπει να διδάσκονται και σε αυτούς τους νέους. Παρακαλώ να το έχετε υπόψη και να το προωθήσετε και αφού φύγω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Πραγματικά θέλω να λάβω υπόψη και την άτυπη εκμάθηση και διδασκαλία. Πολλές δεξιότητες δεν διδάσκονται μόνο στην επίσημη παιδεία, αλλά και σε ανεπίσημους χώρους. Σημαντικό αυτό, αλλά δεν μπορούμε να τα προσμετρήσουμε αυτά. Έχουμε μεγάλη δυσκολία σε αυτό όσον αφορά τον ευρωπαϊκό τομέα της παιδείας. Θέλουμε εκεί να έχουμε αποτελέσματα και βαθμούς στα σχολεία και θέλουμε να έχουμε συγκρίσιμους βαθμούς και επιδόσεις. Στόχος του ευρωπαϊκού τομέα της εκπαίδευσης και αυτόν που αναφέρουμε σε εκθέσεις δεν είναι να ισοπεδώνουμε τα πάντα στα σχολεία, αλλά να έχουμε συγκρίσιμες αποδόσεις, προσμετρήσιμες επιδόσεις. Να πούμε ότι αυτό συγκρίνεται με ένα αποτέλεσμα σε αυτή τη χώρα, διότι έτσι μπορούμε μέσω της σύγκρισης να έχουμε και αποδοχή βαθμών αποτελεσμάτων σε όλη την Ευρώπη στην παιδεία. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε αυτό σήμερα. Όσον αφορά το επίπεδο της παιδείας, δεξιοτήτων και γνώσης διαφέρει τόσο πολύ από χώρα σε χώρα, αυτό πάντα δημιουργεί μεγάλες δυσκολίες αναγνώρισης, ε, απολυτηρίων, αποτελεσμάτων, βαθμών από χώρα σε χώρα σε όλη την Ευρώπη. Το συζητήσαμε αυτό στην ειδική, ειδικού τομεί παιδεία. Το λέγαμε και για συγκεκριμένα πτυχία επαγγελματική εκπαίδευση, η αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών πτυχίων ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη συζήτηση γιατί διαφορετικές χώρες ε, φοβόντουσαν την κατάρρευση της, της εσπερίας γιατί ακριβώς υπάρχουν τόσο μεγάλες διαφορές στα εκπαιδευτικά συστήματα και ιδίω στον τομέα της επαγγελματική κατάρτιση. Οπότε, αν θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευση, όχι μόνο ανώτατη ανώτατης εκπαίδευσης, πρέπει να ενισχυθεί ε, η συγκρισιμότητα μεταξύ των ε, προγραμμάτων σπουδών, των αποτελεσμάτων που επιτυχάνει κανείς και αυτό είναι πολύ σημαντικό και όσον αφορά την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση. Οπότε θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους τομείς <clears throat> χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα μας απασχολήσουν και άλλοι τομείς στους οποίου πρέπει να ενισχυθεί η συγκρισιμότητα. Θα αποτελέσουν σίγουρα όλα αυτά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν την Επιτροπή μας. Στο δρόμο προς τη δημιουργία αυτού του Ευρωπαϊκού Χώρου εκπαίδευση. Αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσει, Σας ευχαριστώ όλους, αγαπητοί συνάδελφοι. Α, ναι, συγγνώμη, ξέχασα να δώσω το λόγο στην, στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή σας που θέτει στην ημερήσια διάταξη αυτό το σημαντικό το θέμα και την Σαβίνα Βεχάιεν την ευχαριστώ για την έκθεσή της. Συμφωνούμε μαζί της. Αυτό είχαμε υπόψη και εμείς όταν ετοιμάσαμε την ετήσια στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2020. Έξοχη γνωμοδότηση. Δύο σημεία μας βρίσκουν ιδιαίτερα συμφώνους. Το πρώτο. Το έγγραφο τονίζει την ανάγκη περισσότερων επενδύσεων σε ποιοτική εκπαίδευση, κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για την πρόθεση οικονομικής αναπτύξεως. Στον τομέα παραγωγικών αυξήσεων και κερδών, λέμε υψηλότερη Παραγωγικότητα και καινοτομία δεν επιτυχάνεται χωρί τι αναγκαίε επενδύσει στην παιδεία και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Και ζητούμε αύξηση των δεξιοτήτων, ψηφιακών δεξιοτήτων και υποστήριξη των εργαζομένων με μαζική αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Αν δίνετε τώρα στον τομέα μακροοικονομική σταθερότητα, το έγγραφο τονίζει την ανάγκη βελτίωση τη ποιότητα των δημοσιονομικών επενδύσεων να προωθηθούν επενδύσεις για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, κυρίως στον τομέα της παιδείας, της απασχόλησης, ότι χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις. Και τέλος, το έγγραφο τονίζει το ρόλο που η παιδεία και η κατάρτιση παίζουν στην προώθηση της δικαιοσύνης, της ισοτιμίας. Στην ετήσια στρατηγική για την ανάπτυξη λέμε ότι χρειάζεται ποιοτική μέρημνα για τα παιδιά και εκπαίδευσή τους, να καλύπτονται όλοι, χρειάζεται ποιοτικό σύστημα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών που εγκαταλείπουν το σχολείο, να βελτιωθεί η ποιότητα της κατάρτισης και να υπάρχει σύγκληση μεταξύ συστημάτων και να υπάρχει επαρκές επίπεδο επενδύσεων για όλα αυτά. Όπως είπαμε στη συζήτηση, το θέμα είναι οι επενδύσεις και όπως είπε και η Μόνικα Σεμέντο, αφορά και διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ισχυρά εργαλεία και για πρόθεση επενδύσεων και για διαθροτική μεταρρύθμιση σε επίπεδο κρατών μελών και δράτω με τις ευκαιρίες να ευχαριστήσω θερμά το Ευρωκοινοβούλιο που προώθησε την ουσιαστική αύξηση του προπολογισμού για το έρασμο για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βοντελάιν, συμφωνεί με αυτό. Και αυτό προωθούμε και στι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Τόσο αφορά διαθωτικές μεταρρυθμίσεις στο μέλλον, θα υπάρχουν δυνατότητες συζήτησης επομένων βημάτων με τον Επίτροπο που θα συζητήσει μαζί σας το διαθρωμένο διάλογο σε ένα μήνα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έρχεται με άδεια χέρια. Προβλέπουμε έκδοση ανακοίνωσης για τον Ευρωπαϊκό τομέα παιδείας, όπου εκεί θα λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα αναφερόμενα σημεία της, ε, του σχεδίου γνωμοδοτήσεως. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνουμε αυτή την δημόσια συζήτηση. Α, καταρχάς να συμπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι 27 Ιανουαρίου στις 12 και παρακαλώ μόνο στα αγγλικά, διότι θα πρέπει να εργαστούμε στα αγγλικά σε αυτό το χαρτοφυλάκιο λόγω χρονικού περιορισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ όλους όσους δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών να αποχωρήσουν τώρα από την αίθουσα και γρήγορα σας παρακαλώ και ήσυχα αν έχετε την καλοσύνη.